κυρία Μαρίν στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Η κυρία Τζίμερ, επικεφαλής της ομάδας GUNGL, κατέθεσε ένα έτοιμο υπεράσπιση των προνομίων και ασύλειών της κυρίας Ελεονόρα Φορέντσα σε σχέση με ένα συμβάν που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαδήλωση στα πλαίσια του G20 στο Αμβούργο. Σύμφωνα με τον κανονισμό, το αίτημα αυτό παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Νομικών